Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω σήμερα στην συνέχεια της ε, συνεδρίασης και χαίρομαι ιδιαίτερος που καλωσορίζω τον κύριο Κοσλόφς, ε, μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου Το θέμα είναι το Euronews. Θα το εξετάσουμε μαζί με τους συναδέλφους της Επιτροπής Ελέγχου του Υπερπολογισμού, αλλά δεν βλέπω κανέναν. Ε, μου είχαν πει ότι κάποιος ε, θα έρθει ή τουλάχιστον τους είχαμε προσκαλέσει. Τον Απρίλιο του 2017 είχαμε κάνει και μια κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Κοντ για την, συντακτική, την εξαρτησία σύνταξης ε, του Euronews και σήμερα ο κύριος ε, Κοσλόφς θα μας παρουσιάσει μια γρήγορη εξέταση της υπόθεσης ε, Euronews το πώς ε, επιτηρεί η Κομισιόν την οικονομική στήριξη στο Euronews για το εάν αυτή είναι αποτελεσματική και με διαφάνεια και αν χρησιμοποιούνται τα κονδύλια σύμφωνα με την εντολή η οποία υπάρχει. Μετά τον κύριο Κοσλόφς ε, θα λάβουν τον λόγο οι βουλευτές ε, για να κάνουν ερωτήσεις ε, και θα απαντήσει ο κύριος Κοσλόφς και η Κομισιόν. Θα του δώσω πρώτα απ' όλα τον λόγο λοιπόν για να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση. 10 με 15 λεπτά. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο της ε, Επιτροπής ε, πρώτα απ' όλα ε, που περιέλαβε το θέμα στη ημερήσια διάταξη και δεύτερον το ότι άνοιξε και την συνεδρίαση αυτή για τους βουλευτές της Επιτροπής ενώ του γιατί είναι σημαντικό αυτό. Μια που είναι η πρώτη μου εμφάνιση στον Κοινοβουλίο θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας, την επανεκλογή σας και να σας ευχηθώ καλή θητεία. Και ως συνήθως το ελεγκτικό συνεδρίο θα σας ε, στήριξει. Δύο λόγια για μένα. Εγώ είμαι μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου στο τέταρτο τμήμα, το οποίο καλύπτει τα οικονομικά, την εσωτερική αγορά και κάποια ζητήματα διοίκησης. Ας έρθουμε τώρα στην εξέταση την ίδια. Πρώτα απ' όλα αφορά την, να ζούμε την φύση του εγγράφου και το πώς εργαζόμαστε εμείς. Οι γρήγορες εξετάσεις αυτές ε, εστιάζουν σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα και συλλέγουν τα σχετικά γεγονότα. Και αν αυτό είναι αναγκαίο μπορεί να περιλάβουν μια ανάλυση για να αντιληφθούμε αυτά τα ζητήματα. Και ε, επίσης θα ήθελα να το τονίσω ότι δεν πρόκειται για έναν πλήρη δημοσιονομικό έλεγχο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε αναλύσει τις σχέσεις μεταξύ Κομισιόν και Euronews και βρήκαμε κάποιες ελλείψεις που θα θέλαμε να αντιμετωπίσει η Κομισιόν επίσης σε όλες τις φάσεις είχαμε εξαιρετική του Euronews, τις δραστηριότητες και τα συστήματα αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά και γαλλικά. η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηριζόταν στο ότι το Euronews ε, παρέχει μια υπηρεσία γενικού συμφέροντος στο, πλαίσιο, στο πεδίο των πληροφοριών. Όμως, ο τρέχον δημοσιονομικός ε, κανονισμός δεν έχει πλέον τέτοια νομική βάση και η Κομισιόν θεωρεί με βάση την απόφαση της του 2010 ότι το Euronews είναι ένας φορέας ο οποίος παρέχει μια δημόσια υπηρεσία στον τομέα της πληροφόρησης. Όμως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν έχουν δώσει έναν τέτοιο ρόλο στο Euronews. Οπότε το Euronews ε, δεν είναι, ή θα μπορούσε να μην είναι προσβάσιμο στους περισσότερους πολίτες ή σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει έλλειψη ενός επίσημου μηχανισμού συντονισμού με την Κομισιόν γιατί οι γενικές διευθύνσεις ε, πέρα από την Γενική Διεύθυνση Connect μπορούν ε, να συνάψουν απευθείας συμβάσεις με το Euronews και η έλλειψη ενός επίσημου μηχανισμού συντονισμού μειώνει την διαφάνεια της οικονομικής ε, στήριξης ε, που δίνεται στο Euronews και ίσως επηρεάζει τη λογοδοσία. Επίσης ε, εξετάσαμε κάποιους εξωτερικούς ελέγχους που είχαν ανατεθεί για να εξεταστούν οι δραστηριότητες του Euronews και κάποιοι σημαντικοί περιορισμοί που είχαν τεθεί από ελέγχους εξάντε για το μηχανισμό μοναδιαίου κόστους δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί αφορούν το σύστημα της χρέους χρόνου και της μέτρησης ε, του ακροατηρίου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ένα κίνδυνο απόκληση μεταξύ μοναδιού κόστους και πραγματικού κόστους. Η Κομισιόν επίσης ε, εισαγαγεί ένα πλαίσιο μέτρησης ε, της απόδοσης για την επίτευξη των στόχων του Euronews. Αυτά υπάρχουν στην Συμφωνία Πλαίσιο. Όμως διαπιστώσαμε ότι η Κομισιόν δεν έχει ε, φτιάξει ένα σύστημα για να επαληθεύσει ε, την λειτουργία αυτή του Euronews και πιο σημαντικό να συνδέσει την απόδοση με την ετήσια απόφαση χρηματοδότησης. Οπότε το Euronews ε, υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στην Κομισιόν αλλά δεν έχουμε δει την σχέση μεταξύ των πληροφοριών αυτών και των ετήσιων αποφάσεων χρηματοδότησης που λαμβάνει η Κομισιόν. Ε, οπότε οι μηχανισμοί ελέγχου απόδοσης ε, πηγαίνουν σε μια βάση ad hoc περισσότερο παρά ενός επισήμου πλαισίου ελέγχου. Οπότε Αυτά Ω μια πολύ σύντομη παρουσίαση της ε, περίπτωσης. Ε, το έγγραφο βεβαίω περιέχει περισσότερα. Σας ε, ευχαριστώ και πάλι λοιπόν που μου δώσατε την ευκαιρία να σα μιλήσω και αναμένω την περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τα εισαγωγικά σας σχόλια, την παρουσίασή σας. Καταρχήν Όποιος θέλει να θέσει ερωτήσεις μεταξύ των μελών και βεβαίως και η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει ερώτηση στον κύριο Κοσλόψ. Θα ξεκινήσουμε όμως με τους, εισηγη... με τους συντονιστές για δύο λεπτά και κατόπιν τα μέλη της Επιτροπής ένα λεπτό. Έχουμε περιορισμένο χρόνο. Χαιρετώ επίσης και την Μόνικα Χολμάιερ, πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμού. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας και θα δώσω το λόγο στην κυρία Ζότροβα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ήταν μια λεπτομερής και εις βάθος παρουσίαση και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Επιτρέψτε μου να κάνω μία σύντομη περίληψη. Αν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρηματοδότηση σε έναν φορέα για δραστηριότητες οι οποίες ουσιαστικά διεκπεραιώνουν μέσω του ιδιωτικού τομέα αυτός ο οργανισμός προηγουμένως ουσιαστικά είχε δεσμευθεί να μην λαμβάνει πλειοψηφικά ή κατά κύριο λόγο χρηματοδότηση από ιδιωτικά ε, κεφάλαια, από ιδιωτικές πηγές. Σήμερα ουσιαστικά αναρωτιόμαστε αν η Euronews πραγματικά προσφέρει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει ιδρυθεί και τις οποίες έχει δεσμευθεί να προσφέρει. Κάνατε μία ανάλυση όσον αφορά τη χρηματοδότηση, όχι όμως όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών. Εντοπίσατε κάποιες αδυναμίες για το πώς οργανώνεται ε, το Euronews όσον αφορά τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο Euronews. Τι συστάσεις όμως έχετε για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, από την ανάλυση που κάνατε μπορείτε να βγάλετε κάποια περαιτέρω συμπεράσματα με τη στήριξη της Επιτροπής ή χωρίς. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αναλύσατε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Euronews. Πρόκειται για έναν σταθμό ο οποίος συμπεριφέρεται, αν θέλετε, σαν ιδιωτικό σταθμός. Πρόκειται για έναν ιδιωτικό φορέα επί του οποίου οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν πραγματικό έλεγχο. Αυτό καταλαβαίνω. Ποιες είναι λοιπόν οι συστάσεις ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυτό. <clears throat> Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω, όπως είπα και στην αρχή της παρουσίασής μου, ότι εμείς εδώ κάνουμε μία έκθεση στην οποία εντοπίζουμε τα πραγματικά γεγονότα και ουσιαστικά τα συμπεράσματά μας απορρέουν από τα γεγονότα και τα στοιχεία που αναλύσαμε. Κατόπιν, οι αρχές, οι αρμόδιες για τα δημοσιονομικά θέματα, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο καλούνται να αποφασίσουν τι κάναμε λοιπόν εμείς. Εμείς ε, εξετάσαμε τη σχέση που υπάρχει σήμερα μεταξύ Euronews και Επιτροπής. Γιατί αυτό μας ζητήθηκε να κάνουμε. Αυτό μας ζήτησε το Κοινοβούλιο. εδώ και πέρα. Εμείς πρέπει να ήδη αποφασίσει να αναλάβουν και τι θέλουν να κάνουν από εδώ και πέρα. Το μοντέλο πάντως που έχει επιλεγεί εδώ και χρόνια για τη στήριξη του Euronews, αν είναι το καλύτερο ή αν υπάρχει και άλλη επιλογή, αυτό είναι άλλο θέμα και θα χρειαστούν άλλες μελέτες. Εμείς στο ελεγκτικό συνέδριο αναλύουμε τώρα την ε, πιθανότητα να αναλύσουμε ξεχωριστά το θέμα των γραμμών του προπολογισμού που απευθύνονται στα οπτικοακουστικά μέσα. Αυτά δεν νομίζω ότι μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι παραπάνω. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας να ακούσουμε την Επιτροπή, να ακούσουμε τι βήματα έχουν αποφασίσει να κάνουν από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ η πρόεδρος της ε, Επιτροπής Προπολογισμού, η Μονικά Χολμάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση που αφορά και την ανάλυση και τα συμπεράσματά σας. Καταλαβαίνω ότι το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των κονδυλίων πάει στο Euronews, έναν σταθμό ο οποίος βρίσκεται σε χέρια ιδιωτών. Υπάρχουν όμως και άλλοι σταθμοί οι οποίοι ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν μπορείτε να μου πείτε αν υπάρχει κάτι στον τομέα των οπτικοακουστικών μέτρων που έχει διαφορετικές συμβάσεις Ξέρουμε πολύ καλά πώς γίνονται αυτές οι συμβάσεις με ανοιχτούς διαχωνισμούς, με πολύ ξεκάθαρες και συγκεκριμένες διαδικασίες. Αυτό που βρίσκω προβληματικό είναι ότι τα κονδύλια παρόν έχετε θέσει και για να δούμε αν λειτουργούν σωστά αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αν υλοποιούνται οι στόχοι ή αν χρειάζεται βελτίωση. Επαναλαμβάνω ότι το ερώτημα είναι αν η καλύτερη προσέγγιση είναι να στηριχθεί ένα. κοινωνικός Και άλλες προσεγγίσεις υπηρεσίας και το ερώτημα είναι αν ναι ή όχι είστε ικανοποιημένοι από την υπηρεσία που παρέχει αυτός ο σταθμός. Επαναλαμβάνω, χρειάζονται ελεγκτικοί μηχανισμοί και σίγουρα μπορεί, αυτό σας το λέω αυτή τη στιγμή μπορώ να το πω ότι χρήζει βελτίωσης ε, ο μηχανισμός αυτός και χρήζει βελτίωσης η υπηρεσία που παρέχεται, η Πέτρα Κάμερβελτ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα συνεχίσω σε σχέση με την τελευταία ερώτηση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και το έγγραφο που μας υποβάλλετε και σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ και χρόνια βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αν κοιτάξει κανείς τον προϋπολογισμό, θυμάμαι ότι είχε γίνει μάχη εδώ στην Επιτροπή μας για να δούμε αν θα, αν χρηματοδοτηθεί μόνο το Euronews ή το Euronet Plus. Και καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέει η Μόνικα Χολμάιερ. Ένας ιδιωτικός φορέας ουσιαστικά αν θέλετε, που έχει συσταθεί, που στηρίζεται ή δεν στηρίζεται από μια συγκεκριμένη κυβέρνηση και πώς ακριβώς συμπεριφέρεται. Αν κοιτάξετε όμως τους κανόνες βάσει των οποίων λειτουργούμε, εδώ υπάρχει θέμα ανταγωνισμού. Και όχι μόνο όσον αφορά την πηγή χρηματοδότησης, από πού δηλαδή ουσιαστικά χρηματοδοτείται, αλλά πιστεύω ότι από τη στιγμή που η κάθε γενική διεύθυνση έχει το δικαίωμα σήμερα να συνάψει δικές της συμβάσεις με την Euronews, καταλαβαίνετε ότι εδώ το σκηνικό μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι προβληματικό, διότι βλέπουμε ότι ποιος τελικά παραγγέλνει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα Παραδείγματο χάρη, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγορά συνάπτει μία συμφωνία, μία σύμβαση με τη Euronews. Και αυτό έχει συνέπειες. Εμείς καλούμεθα μετά να χρηματοδοτήσουμε. Και καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία ολοκληρωμένη εικόνα του τι ακριβώς κάνει, σε ποια έκταση δραστηριοποιείται, πόσα άτομα εργάζονται, πόσοι χρειάζεται, παραδείγματο χάρη, για να διεκπαιρεώσουν από τεχνική απόψεω, πόσα άτομα, αν θέλετε, ουσιαστικά συνεργάζονται και χρηματοδοτούνται στα πλαίσια αυτής της ε, συμβατικής σχέσης. πραγματικά δεν υπάρχει απολύτως καμία αξιολογημέτρηση και απολύτως κανένα στοιχείο το οποίο εδώ να μπορούμε, στο οποίο να μπορούμε να βασιστούμε για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Θα σε ευχαριστώ. Κυρία Κάμεβερτ, καταλαβαίνω με τη γενική ιδέα και συμφωνώ πολύ σωστά τα ερωτήματα που έχετε θέσει. Αλλά επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα του γενικού, του κοινού συμφέροντος, του δημόσιου συμφέροντος. Μέχρι τώρα βασιζόμασταν σε αυτήν την γενική αρχή ότι το Euronews ουσιαστικά εξυπηρετεί σκοπούς δημόσιου συμφέροντος. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν ναι ή όχι αυτό συμβαίνει, συνεχίζει να συμβαίνει. Και αν υπάρχει καλύτερος τρόπος, πιο αποτελεσματικός τρόπος για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Euronews είναι κάτι που δύσκολα μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Αν σήμερα αποφασίσουμε παραδείγματο χάρη να κάνουμε μία μελέτη για να αποτιμήσουμε το κοινό που παρακολουθεί πραγματικά το Euronews, αυτό θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό. Έχουμε λοιπόν πολύ γενικές εκτιμήσεις. Ποιοι είναι οι τηλεθεατές οι οποίοι πραγματικά παρακολουθούν το σταθμό αυτόν. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σήμερα αυτό που συμβαίνει σε πολλά κράτη-μέλη είναι ότι ο σταθμός αυτός δεν υποστηρίζεται από πάρα πολλά κράτη-μέλη. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό πρόβλημα με την, τον αριθμό των τηλεθεατών. Αυτό βεβαίως κατά κάποιο τρόπο εξουδετερώνεται από το θέμα ότι στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το σταθμό αυτό. Υπάρχει και το θέμα της διαφήμισης και από ό,τι μάθαμε θα αυξηθεί η χρηματοδότηση μέσω της διαφήμισης έτσι ώστε να φτάσει ο σταθμός σε μια πιο ισορροπημένη από οικονομικής απόψεως ε, κατάσταση. Σήμερα όμως το 1 τρίτο της χρηματοδότησης του Euronews προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φέγο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η παρουσίαση έρχεται ακριβώ επίκαιρη γιατί συζητάμε τον προπολογισμό. Αυτό που ακούω από την παρουσίασή σα είναι ότι υπάρχουν δύο ισχυρά σημεία. Απ' τη μια η απάντηση στην ανάγκη να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέσο ενημέρωσης, ε, το οποίο να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες Ευρωπαϊκής Ένωσης παντού στην Ευρώπη και ε, ε, σε όλη την Ήπερο η δυνατόν. Και απ' την άλλη υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ Euronews και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, σήμερα ε, δεν έχει επαρκή έλεγχο και σαφήνεια. Από όσα είπατε, κατάλαβα ότι υπάρχει αυτή η διάσταση της εντολής για δημόσια υπηρεσία, δηλαδή δίνουμε ένα ρόλο ε, δημόσιας υπηρεσίας, αλλά δεν έχει δοθεί εντολή. Το να δοθεί λοιπόν μια σαφής εντολή είτε στο Euronews είτε σε κάποιο άλλο κανάλι θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Και δεύτερον, Υπάρχει και ο ε, δημοσιονομικός αντίκτυπος, διότι αυτή η γραμμή προϋπολογισμού ε, βαρύνει ιδιαίτερα τον προϋπολογισμό μας και θα πρέπει να το παρακολουθούμε στενά γιατί δημοσιοποιείται και όλο αυτό το θέμα. Και αυτή η γραμμή ξεκίνησε γιατί υπήρχαν και ε, προκλήσεις όσον αφορά ε, τον, ε, ε, τη μετάφραση. Πρέπει όμως να παρακολουθήσουμε και τι γίνεται για τη σαφή ε, χρήση αυτών των κονδυλίων. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το Euronews ε, σίγουρα δεν είναι το τέλειο, αλλά οι πληροφορίες που διαθέτουμε και που διευκρινίζετε και εσείς στην έκθεσή σας ε, καταδεικνύουν ότι υπάρχει και ανεξάρτητη δημοσιογραφία, υπάρχει και μία ποιότητα την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, αλλά φυσικά τίθεται το θέμα ε, που έθεσε και η κυρία Κάμερ-Εύερτ ε, ε, των τηλεθεατών και του αριθμού των τηλεθεατών και θα πρέπει να γίνουν και πλήρης έλεγχοι για να γνωρίζουμε και τι θέλουμε εμείς ως ευρωπαϊκό μέσο ενημέρωσης και να δώσουμε ένα τέλος ίσως σε αυτή την εταιρική σχέση με το Euronews αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι αυτό που θέλουμε. Εγώ θα ήθελα να δω και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι μπορούμε να βελτιώσουμε σε αυτή τη σχέση από πλευράς αποτελεσματικότητας, αλλά ίσως και κάποιες εναλλακτικέ λύσεις, εάν ε, ολοκληρωθεί αυτή η σχέση, διακοπή μάλλον. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Νομίζω ότι αν ε, πάμε στη σύσταση της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Euronews και η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Euronews ε, αποτελούσε προτεραιότητα του αρμόδιου επιτρόπου, ε, της Επιτρόπου Μαρίσα Γκαμπριέλ. Και για να επιστρέψω και στο θέμα της αποτελεσματικότητας και του αριθμού των τηλεθεατών, της θεαματικότητας, να υπενθυμίσω ότι το Euronews έκανε κάποιες βελτιώσεις στο επιχειρηματικό του μοντέλο. Αντί για την κατάσταση που είχαμε στο παρελθόν, όπου υπήρχε ένα βίντεο το οποίο μεταφραζόταν σε αρκετές γλώσσες, Τώρα για να αυξηθεί η θεαματικότητα και να έχουμε μια προσέγγιση η οποία θα είναι πιο πολύ στα μέτρα του κοινού, το Euronews δημιουργεί διαφορετικά βίντεο σε διαφορετικές γλώσσες για το ίδιο θέμα. προσαρμόζουν ουσιαστικά τις πληροφορίες ε, στη γεωγραφική περιοχή στην οποία ε, μεταδίδεται ε, το κανάλι αυτός είναι ένας τρόπος να αυξηθεί η θεματικότητα. Τώρα, το κατά πόσον βοήθησε ή όχι, δεν το αναλύσαμε εμείς. Ίσως οι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαν ε, να απαντήσουν. Και επίσης, όπως σας είπα, ένα από τα συμπεράσματά μας είναι ότι δεν έχουμε δει άμεση σχέση μεταξύ των επιχειρησιακών πληροφοριών της Euronews ε, για τις επιδόσεις τους και τις ε, αποφάσεις που λαμβάνονται για την για τις ετήσιες ε, χρηματοδοτήσεις. Αυτό είναι ίσως κάτι το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί καταρχάς και από εκεί και πέρα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να μπορέσουμε να κρίνουμε κατά πόσον η υπογραφή της ε, συμφωνίας ε, αιτιολογείται ή όχι. Ευχαριστώ. Η κυρία Χέρμπουν. Ζητήσατε το λόγο. Merci. Ευχαριστώ. Εγώ θα συμφωνήσω απολύτως με την προλαλήσασα. Να πω κι εγώ κάποια πράγματα. Εγώ αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι, σε σχέση και με αυτά που διάβασα, είναι ότι αυτή τη στιγμή ε, υπάρχουν ε, ελλείψεις ε, από πλευράς Euronews, αλλά και κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να ε, προσάψουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέμε στα γαλλικά ότι δεν μπορούμε να πετάξουμε το μωρό μαζί με τα απόνερα. Εγώ νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το σώσουμε το βρέφος. υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις οι οποίες έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης διάβασα τις διάφορες απόψεις και διάβασα ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αυτή η οποία προέτρεψε το Euronews να βρει και άλλους επενδυτές. Το ερώτημα ήταν κατά πόσον έχει πλαισιωθεί καταλήλως. Έχει ζητηθεί επισήμως ε, να είναι μόνο Ευρωπαίοι επενδυτές ή θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε και ε, επενδυτέ εκτός Ευρωπαϊκή Ένωσης. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και πλεονέκτημα, διότι ε, έχουμε και διεθνές ε, ε, κοινό και ε, κάποιους οι οποίοι δεν θα είχαν δει ποτέ το κανάλι αυτό αν ήταν αμυγός ευρωπαϊκό. Επιπλέον, εγώ εκπλήσωμαι και λίγο, διότι Προηγουμένως λέγαμε όλοι ότι εφαρμόστηκαν κάποια ε, μέσα για τον έλεγχο, αλλά τελικά ο έλεγχος δεν έγινε. Και θα ήθελα να ξέρω γιατί δεν έγινε ο έλεγχος. Ακούστηκε επίσης ε, και ότι ίσως θα έπρεπε να ε, πάει στο Euronet ένα τμήμα της χρηματοδότησης και εδώ τίθεται το ίδιο ερώτημα. Εάν δεν καταλήξουμε σε συμπέρασμα για το τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δεν έκανε ή τι δεν έκανε και το Euronews, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Άντερσον, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά παρακολουθούμε τη σειρά των ε, ομιλητών σε σχέση με το μέγεθος των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Άντερσον έχει το λόγο. Καλημέρα, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα του Euronews είναι προβληματικό. Αυτό το ακούμε από όλε τι πλευρέ. Χρειάζεται σίγουρα μια πιο βαθιά ανάλυση των δυσκολιών και των ε, προβλημάτων. Ακούσαμε και την πρόεδρο τη Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προλίγμου. Αυτό που όμως διαπιστώνουμε είναι ότι το Euronews δεν είναι ένα κανονικό ε, ένας κανονικός οργανισμός ε, τηλεοπτικός. Πρόκειται για κάτι που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό και θα πρέπει να έχει διαφορετικούς σκοπούς. Όσον αφορά τη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνουμε ότι εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη αποστολή να αναλύονται τα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ενδεχομένως στην ζωή των κρατών μελών και των Ευρωπαίων πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν εδώ να ξαναδούμε αυτούς τους στόχους, να δούμε παραδείγματο χάρη θέματα ποιότητας, θέματα συντακτικής ουδετερότητας κτλ. Χρειάζεται λοιπόν να ξαναδούμε τι υπηρεσία παρέχεται βάσει αυτού του συμβολέου, βάσει αυτής της σύμβασης, βλέπουμε ότι σήμερα οκτώ διαφορετικές γενικές διευθύνσεις έχουν συνάψει χωρίς συντονισμό και χωρίς έλεγχο από κανένα συμβάσεις με τον σταθμό Euronews. Και ουσιαστικά μόνο το 15% της ιδιοκτησίας αυτού του σταθμού ανήκουν πραγματικά σε ευρωπαϊκά χέρια. Αν κοιτάξει κανείς τον προϋπολογισμό, διαπιστώνει ότι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος θα πρέπει να ενημερωθεί για το τι ακριβώς συμβαίνει. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει και αναφέρεται στα μονοπόλια, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στο κατά πόσο αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Όμως για μένα το συμπέρασμα είναι ότι σε καμία περίπτωση ένας τέτοιος τηλεοπτικός σταθμός, ένας σταθμός ε, τέτοιου είδους δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται σε καμία περίπτωση και σε κανένα βαθμό από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να ελέγξουμε ακριβώς τι συμβαίνει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Euronews και θα πρέπει να γίνει εδώ μία εις βάθος ανάλυση από μέρους του ελεκτικού συνεδρίου. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι γραμμές, οι κατευθύνσεις, η συντακτική, αν θέλετε, πολιτική αυτού του σταθμού και την ίδια ώρα να δούμε πώς οι Ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται και έχουν πρόσβαση στο Euronews Ποιος είναι ο ρόλος του Euronews σε θέματα που αφορούν παραδείγματος χάρη το Brexit. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα θέματα αυτά που απασχολούν αυτόν τον σταθμό. Και νομίζω ότι όλα αυτά που αναφέρουμε εδώ είναι θέματα που θα άξιζαν μια εις βάθος συζήτηση. Ο κύριο Κοσλό, ευχαριστώ. Νομίζω ότι και αυτό και τα άλλα σχόλια ήταν γενική φύσεω σχόλια και νομίζω ότι εκφράσατε τις απόψεις σας βάσει και των πληροφοριών που σας δώσαμε, αλλά και βάσει ε, άλλων πληροφοριών. Εμείς εξετάσαμε κάποια στοιχεία από το πρίσμα τι ε, σχέσεις και τη στήριξη και τη χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, αλλά θέλουμε να τα αναλύσουμε και να δώσουμε πληροφορίε για το κατά πόσον είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείται αυτή η σχέση και ε, πώς υποβάλλονται οι εκθέσεις για τη σχέση αυτή. Και το πρώτο βήμα θα ήταν να δούμε εάν και κατά πόσον ε, αυτή η σχέση θα μπορούσε να βελτιωθεί. Μέχρι αυτού του σημείου μπορώ εγώ να σχολιάσω ως μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου επί του ζητήματος. Ευχαριστώ. Ja, Σας ευχαριστώ. κύριος Κιζιγιούρεκ, τελευταίος συντονιστής. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι διάβασα την έκθεση και είδα κάπου εκεί στη σελίδα 9 κάποιο παρατηρητήριο Σερβατόριο Τυπάβια, ένα ανεξάρτητο εξωτερικό Ινστιτούτο Ανάλυσης ε, των Επικοινωνιών που λέει ότι το Euronews ε, είναι προσιλωμένο στην ακαιρεότητα και την αμεροληψία, δεν υπονομεύθηκε ποτέ η άποψη των δημοσιογράφων κτλ. Δηλαδή ε, εδώ πέρα μου λέει ότι τα πράγματα πάνε καλά από την δημοσιογραφική σκοπιά. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι δεν πρέπει να περικοπούν οι διάφορες γλώσσες ε, για να είναι προσβάσιμα αυτά τα προγράμματα. Τώρα, το Euronews ε, Ε, κατά την άποψή μου βοηθάει πάρα πολύ για να υπάρξει ένας κοινός δημόσιος χώρος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ το κοινό το βλέπω κάπως διαφορετικά από το CNN, οπότε υπ' αυτήν την έννοια είναι πολύ σημαντικά αυτά τα προγράμματα. Τώρα, ε, λέτε στην έκθεση πως υπάρχουν κάποια ελλείμματα. δεν μπορώ από αυτό να εκφράσω άποψη, αλλά θα ήθελα ε, να ακούσω και την άποψη του Euronews ε, επί της έκθεσης αυτής ε, ε, απάντησε το Euronews σε αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να ακούσω και τα δικά τους επιχειρήματα, γιατί προφανώς τα πράγματα από δημοσιογραφική σκοπιά δεν είναι άσχημα και κατά βάση αυτό έχει σημασία. Και αυτή είναι μια ε, τοποθέτηση παρά μια ερώτηση μάλλον. Θα δώσουμε την ευκαιρία και στην Κομισιό να τοποθετηθεί που αναφέρθηκε πολλές φορές. Σήμερα δεν είχε προβλεφθεί να ακούσουμε το Euronews. Σήμερα έχουμε την επίσημη έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και την τοποθέτηση της Κομισιόν. Οπωσδήποτε το θέμα θα μας απασχολήσει τους επόμενους ε, μήνες και εβδομάδες. Στο πλαίσιο του και του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγραμματισμού. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει ότι ε, το Euronews ε, μεταδίδει τώρα τις απόψεις της ε, Κομισιόν, αν το δει κανείς. Οπωσδήποτε στη συμβάσεις υπάρχει και η ανεξαρτησία από την Κομισιόν ε, που χρηματοδοτεί και νομίζω ότι δεν υπάρχει άμεση επιρροή της Κομισιόν στην σύνταξη. Λοιπόν, ούτως ή άλλως δεν ξεκαθαρίζουμε αυτό σήμερα αλλά το εάν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ελέγχου και αν λειτουργεί σωστά, εάν γίνονται οι έλεγχοι. Αυτό είναι κατ' ουσίαν ε, το περιεχόμενο της έκθεσης, οπότε θα ήθελα σήμερα να περιοριστούμε σε αυτά τα οποία μας απασχολούν και τα συμπεράσματα που βγάζει ο καθένας ε, νομίζω είναι για μια άλλη στιγμή. Έχω μία ερώτηση εγώ για το θέμα των ελεγκτικών μηχανισμών, δηλαδή το πώς υπάρχει αυτή η πληροφόρηση μεταξύ του σταθμού και της ε, Κομισιόν. Δεν κάνει τίποτα η Κομισιόν. Τι γίνεται. Πώς ε, βλέπετε αυτά τα οποία κάνει η Κομισιόν στο πλαίσιο της συμφωνίας ε, με την Κομισιόν είναι αμέλεια του Euronews ή είναι θέμα του εάν ασχολείται καν η Κομισιόν με την συμφωνία αυτή. Αυτή είναι η δική μου ερώτηση και να κάνω και ένα σχολείο Είναι νομίζω σημαντικό ότι και από την Ευρωπαϊκή Σκοπιά να έχουμε πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από μια ευρωπαϊκή οπτική γωνία γιατί η εθνική τηλεοπτικοί σταθμοί δεν το κάνουν ή το κάνουν πάντα από μια εθνική σκοπιά. Καλό είναι να υπάρχει και ένας κοινό ευρωπαϊκός χώρος ε, πληροφόρησης. Ε, τώρα το ποιος θα το κάνει αυτό τελικά εντάξει είναι κάτι το οποίο παραμένει ανοιχτό. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, πρόσφορες στον τομέα αυτών και συνεργασίες. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τους ή άλλους και τους επόμενους ε, μήνες όταν θα δούμε την κατεύθυνση του προγράμματος. Κύριε Κοσλόφς, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, στα συμπεράσματα αυτά βρήκαμε ότι στο είναι συμφωνία πλαίσιο υπάρχουν ε, διάφοροι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες και το Euronews δίνει τακτικά αυτές τις ε, πληροφορίες στην Κομισιόν. Στο επιχειρησιακό επίπεδο η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ε, Euronews και Κομισιόν λειτουργεί καλά. Εκεί όπου βρήκαμε κάποιες ε, δυσκολίες είναι στο πώς η Κομισιόν χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες. στην απόφαση της ε, για την ετήσια χρηματοδότηση. Το εάν αξιολογείται ε, η πληροφορία αυτή στην περαιτέρω λήψη αποφάσεων. Αυτό τονίζουμε σε ένα από τα συμπεράσματά μας. Ότι ίσως χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες από την Κομισιόν και πιθανώς ε, βελτιώσεις. Και για να αναφερθώ και στην ε, ανεξαρτησία. Πράγματι, ένα από τα συμπεράσματά μας είναι πως διάφορες ε, ε, ανεξάρτητες εκθέσεις από το Σερβατόριο τη Πάβια δεν βρήκαν σοβαρές και καθόλου παραβιάσεις της ανεξαρτησίας της δημοσιογραφικής. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι οι μελέτες αυτές χρηματοδοτούνται από το ίδιο το Euronews βέβαια. Κατ' οποίο δεν σημαίνει από μόνο του ότι είναι λιγότερο έγκυρες. Μια βελτίωση θα μπορούσε να είναι ε, τις μελέτες αυτές να τις αναθέτει η Κομισιόν και έτσι ε, θα είχαμε ένα αυξημένο βαθμό ανεξαρτησίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις έχω. Ένα λεπτό παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. κύριος Φούρλας πρώτα και μετά κυρία Κάμερεβερτ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπε μια καλή συνάδελφος προηγουμένως ότι δεν πετάμε το μωρό μαζί με τα απόνερα. Εγώ δεν βλέπω εδώ το μωρό σήμερα για να ακούσει αυτά που λέμε και να φέρουμε στο Euronews. Αν έχει καλεστεί και δεν έχει έρθει εδώ το Euronews, παρόλο που δεν οφείλει να μιλήσει σήμερα, το θεωρώ απαξίωση για την επιτροπή στην οποία είμαστε σήμερα εδώ. Ε, εποπτικό μηχανισμό. Είπατε εσεί ο ίδιο ότι δεν υπάρχει επαρκή εποπτικό μηχανισμό. Άρα, αυτό που εγώ συμπεραίνω ω νέο ευρωβουλευτή είναι ότι χρηματοδοτούμε το Euronews, αλλά δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Είμαι δημοσιογράφο και δεν δεχόμουν ποτέ να παρέμβει κάποιο στην ανεξαρτησία μου. Άρα το Euronews καλά κάνει και έχει την ανεξαρτησία του. Κάποια θέματα όμω, επειδή είπατε ότι οφείλει να υπηρετεί την ευρωπαϊκή σκοπιά. Και θέτω ένα παράδειγμα. Επιβάλλεται να γίνονται σεβαστά τα τοπονύμια των κρατών μελών όπω τα ορίζει το κράτο μέλο. Το Euronews πάρα πολλέ φορέ αναφερόταν στην κατεχόμενη Κύπρο με τα παράνομα, αν θέλετε, τοπονύμια. Όταν τέθηκε αυτό το θέμα από συναδέλφου, η απάντηση ξέρετε ποια ήταν. Ξέρετε, το Euronews είναι ιδιωτικό οργανισμό. Αν αυτή η απάντηση θα λαμβάνουμε κάθε φορά που θέτουμε κάτι, θα πρέπει να δούμε και το θέμα τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο με ενοχλεί εμένα είναι ότι από ό,τι φαίνεται είναι αυτοματισμός εδώ πέρα. Η Κομισιόν δηλαδή δίνει τα λεφτά ανεξαρτήτως ε, του τι ε, λέει η έκθεση και του αν υπάρχει κάποιος ε, έλεγχος. Έτσι, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Το βασικό ερώτημα λοιπόν εδώ πέρα που πρέπει να θέσουμε είναι το εξής. Μήπως υπάρχει μια άλλη καλύτερη προσφορά που θα μπορούσε να υλοποιήσει με καλύτερο τρόπο αυτό το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον καλύτερα από το Euronews. Ε, Παραδείγματο χάρη ε, στο Facebook υπάρχει ένα πρόγραμμα της Deutsche Welle συνεργασία με την ε, France Media που έχει πολλαπλάσιους θεατές από το Euronews. Λοιπόν, το ερώτημα είναι ακριβώς με ποιον τρόπο θα πετύχουμε καλύτερα τον σκοπό μας. Και θα μπορούσαμε έτσι να χρηματοδοτήσουμε διάφορες πιθανότητες. Σας ευχαριστώ. Κύριος Νίνας. Κοιτάξτε. Πρέπει να είναι ανεξάρτητο αυτό το οποίο μεταδίδει το Euronews από την χρηματοδότηση. Αλλιώς θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Έχω όμως ε, μια άλλη ερώτηση. η πώληση του 85% ε, πώς συνέβη και δεν ξέρω μπορεί να αναστραφεί για να επανέλθουμε στο προηγούμενο ε, status quo γιατί αν δεν είναι ιδιωτικό δεν θα έχουμε και τα προβλήματα αυτά. παρόλα αυτά το Euronews είναι ένας ε, σταθμός ο οποίος ε, είναι εκτός εποχής πλέον. Δηλαδή η αναλογική τηλεόραση προς, που πηγαίνει προς μία κατεύθυνση μόνο έχει πεθάνει εδώ και δεκαετίες. Πρέπει να δούμε κάτι το οποίο θα είναι πιο σύγχρονο κάπως. Ένα, μια ευρωπαϊκή ραδιοτηλεόραση. Αυτό είναι το ένα και το άλλο, όπως σας είπα, μπορούμε να τον ξαναγοράσουμε το σταθμό με κάποιον τρόπο. Λοιπόν, έχετε τον λόγο και μετά θα δώσω τον λόγο στην Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Στο εγγραφό μας αναφέρουμε το πώς ε, έχει η ιδιοκτησία του σταθμού. Αρχικά ήταν ε, 100% ιδιοκτησία των ευρωπαϊκών ε, κρατικών ε, ραδιοσταθμών. Σε κάποια φάση, για λόγους τους οποίους εγώ δεν γνωρίζω, ως μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, ε, δεν υπήρχε πλέον η όρεξη των δημοσίων ραδιοτηλεοράσεων να συνεχίσουν να επενδύουν και να είναι μέτοχοι στο Euronews και να στηρίζουν το κανάλι αυτό. και η Κομισιόν μετά θεώρησε ότι ο μόνος τρόπος ε, ήταν να βρεθούν ε, ιδιώτες επενδυτές και έτσι έγινε. Πρώτα η εταιρεία αυτή, η Amgen, μια εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο, η ιδιοκτησία ενός Αιγυπτίου ε, και μετά το NBC. Ε, καθένας από αυτούς ε, δημιέφερε κάποια νέα χαρακτηριστικά το NBC παραδείγματος χάρη ε, σήμανε την ψηφιοποίηση κάποιων γλωσσών και δεύτερον την ανάπτυξη ενό πιο ανταγωνιστικού αγγλόφωνου καναλιού με περισσότερους δημοσιογράφους επιτόπου κτλ. Αυτό δηλαδή για να στηρίξω αυτό το οποίο είπα, ότι οι ιδιώτες επενδυτές ε, επέφεραν κάποιες βελτιώσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο. Θα έλεγα ότι το έκανα πιο ανταγωνιστικό το Euronews, αλλά προφανώς αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το χρηματοδοτήσει ή όχι. Αντικειμενικά έγιναν πιο ανταγωνιστικοί. Το ερώτημα τώρα είναι αν ε, θεωρούμε ότι το γενικό δημόσιο συμφέρον μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα από το Euronews με άλλον τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα χαιρετήσουμε τώρα την Επιτροπή, τον κύριο Αγουαμόντε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Πολλά σημεία αναλύθηκαν και εγώ θα ξεκινήσω αποσαφηνίζοντας την οικονομική σχέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Euronews. Μέχρι το, μάλλον από το 1993 ξεκινάμε. Αρχικά ο προϋπολογισμός ήταν 2 με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Από το 2010 υπάρχει ε, μία σύμβαση πλαίσιο και από το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά δίνει 18 εκατομμύρια στο Euronews το χρόνο για το σύνολο των ε, προγραμμάτων Κάτι που ο κύριος Κόσλοφ ανέφερε στο τέλος είναι καθοριστικό, δηλαδή ο ενθουσιασμός του κοινού, αν θέλετε. Το Euronews δημιουργήθηκε με την συνεργασία πολλών ευρωπαϊκών φορέων και βεβαίως ξεκίνησε σαν ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα η οικονομική δέσμευση όλων αυτών σιγά σιγά όμως αποδυναμώθηκε. Και αν ήθελε να επιβιώσει το Euronews έπρεπε να βρεθεί εξωτερική χρηματοδότηση. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης. Γι' αυτό ακριβώς και ο Επίτροπος ε, Έτιγκερ και Γκάμπριελ έπρεπε, αν θέλετε, να στηρίξουν το Euronews και να βρει ένα υγιές επιχειρηματικό μοντέλο, να επιβιώσει. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ξεκάθαρο από την έκθεση αυτή. Στην αρχή της έκθεσης διαβάζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε το σταθμό Euronews έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, να ε, προσελκύσει νέα χρηματοδότηση και να στηριχτεί σε ένα υγιές επιχειρηματικό μοντέλο. Και αυτό το έκαναν και οι δύο αρμόδιοι επίτροποι. Πολλά έχουν ακουστεί όσον αφορά τον έλεγχο. Βεβαίως, ο έλεγχος μπορεί να είναι καλύτερος. και πραγματικά ε, όλα τα πράγματα μπορεί να γίνουν καλύτερα, η έλεγχη μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες διαδικασίες και υπάρχει το πλαίσιο το οποίο προβλέπει κάθε δύο χρόνια έναν πολύ σημαντικό εξωτερικό έλεγχο. Κάθε χρόνο δε γίνεται ο εσωτερικός έλεγχος. Κάθε χρόνο. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Η τελευταία εξωτερική αξιολόγηση που έκανε η εταιρεία Deloitte το 18 έφτασε στο συμπέρασμα ότι ο σταθμός Euronews είναι χαμηλού κόστους αποτελεσματικός οργανισμός και ότι υλοποιεί με αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά θέματα λογοδοσίας, διαφάνειας, Βεβαίως η έκθεση αυτή εντόπισε κάποιες αδυναμίες όσον αφορά την συντακτική πολιτική και κάτι που εμείς το αναλάβαμε. Ξεκινήσαμε με ένα σχέδιο δράσης με σκοπό να γίνουν συνεδριάσεις με όλες αυτές τις ε, γενικές διευθύνσεις οι οποίες έχουν συνάψει συμβάσεις και ε, έχουν ε, σχέση με το Euronews για όλες αυτές, όλα αυτά τα προγράμματα έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και έλεγχος για να απαντήσω στο ερώτημα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτήν την έκθεση. Κάποιες από τις δράσεις θα πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικές και πιο ε, οικονομικές. Δηλαδή, θέσαμε ερωτήσεις πολύ συγκεκριμένα για τις περικοπές κόστους και η μετατροπή του καναλιού σε ένα ψηφιακό κανάλι σίγουρα θα απελευθέρωνε περισσότερα κονδύλια για περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η βελτίωση των ελέγχων τώρα. Αυτό λέτε στην έκθεση. Λέτε ότι υπάρχουν ε, οι μηχανισμοί ελέγχου, λέει ότι δεν χρησιμοποιούνται συστηματικά και ότι μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους. Υπάρχουν τρόποι να υπάρξει πιο συστηματικός έλεγχος, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας. Στο σχέδιο δράσης μας ασχοληθήκαμε και με το παρατηρητήριο της, ε, της ε, Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο οργανισμό που δεν βρήκε απολύτως τίποτα το οποίο να φαίνεται σαν ε, λάθος διαδικασία ή ανομαλία στη λειτουργία. Θα τους ξανασυναντήσουμε όμως, το παρατηρήτιο αυτό, την επόμενη εβδομάδα ο επιχειρηματίας, ο Αιγύπτιος, ο κύριος Σαουίρη, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή τον έλεγχο του Euronews, τηρεί και έχει προσυπογράψει την σύμβαση για την συντακτική ανεξαρτησία του Euronews. Υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες όσον αφορά διαμαρτυρίες, προσφυγές για θέματα που αφορούν το περιεχόμενο. Πολλά λοιπόν γίνονται. Βεβαίως έχετε δίκιο, μπορούμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες. Αλλά πραγματικά ε, μην ε, θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι να μιλήσω ακόμα δύο λεπτά, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχει ένα νομικό θέμα στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που αφορά τη νομική βάση. Διαφωνώ με το ελεγκτικό συνέδριο γιατί υπάρχει το νέο άρθρο 180 παράγραφος Β και το 194 στο δημοσιονομικό κανονισμό που αποτελεί ουσιαστικά τη νομική βάση για τη χρηματοδότηση του Euronews. Μπορώ να σας το εξηγήσω και μάλιστα το αρμόδιο τμήμα για τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ελέγξει ακριβώς αυτή τη νομική βάση, βάση της οποίας χρηματοδοτείται το Euronews το λογιστικό σύστημα στο Euronews δεν είναι αρκετά αναλυτικό έτσι ώστε να συμπεριλάβει κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στον λογιστικό έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει αρκετά αναλυτικό σύστημα στα λογιστικά του Euronews για να δοθούν κάποια στοιχεία, αλλά ότι αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο και μάλιστα μας υποσχέθηκαν ότι από το Φεβρουάριο του επόμενου έτους θα θεσπίσουν ένα νέο σύστημα, θα υιοθετήσουν ένα νέο λογιστικό σύστημα το οποίο θα είναι αρκετά αναλυτικό για να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές που ζήτησε ο ελεγκτής. ...5,3 εκατομμύρια σε 16 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολούθησαν το 2018 το Euronews. Αναρωτιέμαι εάν μπορούμε να λάβουμε αυτό το action plan για το οποίο μιλάτε. Να δούμε τι γράφει και τι εφαρμόζεται εκεί πέρα. Και για την Επιτροπή του Προπολογισμού αυτά τα έγγραφα του εξωτερικού ελέγχου. Τι έχει να πει η Deloitte για αυτά τα ζητήματα. Το δεύτερο ερώτημα. είναι μεταξύ η κατάσταση έχει αλλάξει από όταν ξεκίνησε η οικονομική ενίσχυση του Euronews. Υπήρχε τότε αυτός ο συνεταιρισμός δημοσίων ραδιοτηλεοράσεων που έφτιαξαν αυτόν τον ευρωπαϊκό σταθμό, αλλά σήμερα έχουμε πάρα πολλά πιλωτικά σχέδια με ευρωπαϊκή δημοσιογραφία από πολλούς και διάφορους ε, στον ακουστικό τομέα, στο διαδίκτυο Οπότε σε ποιο βαθμό μπορούμε πλέον να έχουμε αποκλειστικά τη χρηματοδότηση ενός σταθμού ο οποίος δεν είναι πλέον και κρατικός. Η απάντηση στην ερώτησή σας ε, για το σχέδιο δράσης είναι κάτι το οποίο εκπονήθηκε από εμά μετά από τον έλεγχο προκειμένου για να απαντήσουμε, να απαντήσουμε στις συστάσεις του ελέγχου, δηλαδή να βελτιώσουμε τους υφιστάμενους ελέγχους. Ε, πολύ ευχαρίστω να σας το στείλω όταν θα επιστρέψει στο γραφείο μου. Στο παρατηρητήριο της Παβία ε, θα έρθω σε επαφή μαζί τους τις επόμενες μέρες και θα δούμε κατά πόσον ε, είναι απαραίτητο να γίνει ένας περαιτέρω ανεξάρτητος έλεγχος αυτή τη φορά, ο οποίος ε, θα πληρωθεί από το, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για άλλη μια φορά, αν επιμένετε ούτως ή άλλως θα γίνει, αλλά για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια και πραγματικά έχουμε ασχοληθεί πολύ καιρό με το Euronews, ε, το γεγονός ότι υπάρχουν δημόσιες τηλεοράσεις οι οποίες ακόμα ε, συμμετέχουν στο Euronews και δεν είχαν καμία ένδειξη ότι ε, η δημοσιογραφική ε, πλευρά της, του Euronews δεν είναι ανεξάρτητη. Κανείς δεν αμφισβητεί την ανεξαρτησία του Euronews. Ελήφθη κάποια στιγμή μια πολιτική απόφαση που περιλαμβανόταν στην ε, ε, επιστολή της εντολής. Εγώ απλώς σημειώνω ότι η επιθυμία σας είναι η νέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τι μπορεί να αντέξει η αγορά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάμερεβερ και κυρία Χολμάγερ σαν επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Η κυρία Κάμερεβερ πρώτα. Ευχαριστώ. Άλλη μια ερώτηση θέλω να κάνω, κυρίως ε, μετά την ερώτηση που έκανε η Πρόεδρος. Τι άλλες δυνατότητες έχουμε στην Ευρώπη που μπορούμε να στηρίξουμε. Έχετε σκεφτεί συγκεκριμένα εσείς σαν Επιτροπή και θα συνεισφέρετε έτσι ώστε να υπάρξει περισσότερη πολυμορφία περισσότερη, αν θέλετε, δυνατότητα επιλογής. Αυτό είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς δηλαδή θα δαπανηθούν τα ποσά αυτά που προβλέπονται σε αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού για αυτό το τομέα. Έχετε σκεφτεί στην Επιτροπή κάτι τέτοιο ή περιμένετε μέχρι να έχετε νέα πρόεδρο στην Επιτροπή για να σας δώσει οδηγίες. Πώς θα πετύχουμε περισσότερη πολυμορφία, περισσότερη επιλογή. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Και πραγματικά πώς θα πετύχουμε περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ευρωπαϊκές πληροφορίες. Κυρία Χολμάιερ, εγώ βεβαίως ε, Καταλαβαίνω ότι αυτές οι δυνατότητες σύμβασης υπάρχουν και επιτρέπεται να δίνονται με αυτό τον τρόπο. Η ερώτηση μου είναι, θα περιοριστούμε σε ένα μοναδικό μέσο το οποίο θα στηρίζουμε και θα χρηματοδοτούμε. Εδώ βλέπετε ότι ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι αγοράζουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο σε έναν σταθμό και ουσιαστικά βάζουμε το δικό μας περιεχόμενο και προσπαθούμε να το διαδώσουμε στις χώρες της Ευρώπης. Υπάρχει και μία άλλη όμως εναλλακτική. Παίρνουμε πολλά μέσα, πολλές δυνατότητες, πολλά δίκτυα και κανάλια και ουσιαστικά δίνουμε μία συγκεκριμένη ε, κατεύθυνση και σε αυτή την περίπτωση ελέγχουμε και την συντακτική γραμμή αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά τίθεται υπό την αιγίδα της εκάστοτε σύνταξης. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ε, μου φαίνεται ότι από νομικής απόψεως υπάρχουν κάποιες ε, δυσκολίες. Είναι λίγο προβληματικό ε, δεν είναι δηλαδή το ερώτημα μόνο αν τα κονδύλια δαπανώνται με σωστό ή λάθος τρόπο, με κανονικό, με ομαλό τρόπο από δημοσιονομικής απόψης. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άλλα κανάλια και άλλοι φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να στηριχτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ζητήσουμε εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με την Επιτροπή ο τρόπος που έχει συναυθεί αυτή η σύμβαση για μένα είναι προβληματική. Δεν πρόκειται για κάτι απλό ότι εμείς συνάπτουμε μια συμφωνία και ε, χρησιμοποιούμε μια δυνατότητα για να μεταφέρουμε συγκεκριμένες ιδέες και πληροφορίες. Εδώ πρόκειται για θέματα που άπτονται και της ε, ελευθερίας έκφρασης και πολλών άλλων πραγμάτων. Υπάρχουν νομικά προβλήματα, και υπάρχουν και θέματα χρηματοδότησης. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Βεβαίως έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Κυρία Φεράν και ο κύριος Κοσλός και ο κύριος Αμπαμόντ μπορούν να ξαναπάρουν το λόγο. Πολύ σύντομα όμως παρακαλώ, γιατί έχουμε και άλλο ένα θέμα πριν τη συνάντηση των συντονιστών. Η κυρία Φεγό, σύντομα και πέρα για το συγκεκριμένο θέμα. Μιλάω και εγώ για την πολυμορφία. Πρέπει να προσέξουμε γιατί όσον αφορά τα μέσα, καταλαβαίνετε χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη δύναμη, ένα συγκεκριμένο μέγεθος για να μπορεί να υπάρξει ευρεία διάδοση και δυνατότητες μετάφρασης. Αυτό προϋποθέτει μια δύναμη, ένα βάρος και μια επιρροή. Ευχαριστώ. Κύριε Κοσλός και μετά ο κύριος Αμπραμόντ. Oh. Ναι, νομίζω εξ ονόματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση, η οποία ήταν ιδιαίτερα ζωηρή, όπως περίμενα άλλωστε. Και χαίρομαι που η δική μας η αναθεώρηση που έγινε με την ταχύοδό σας προσέφερε και δυνατότητες να σκεφτείτε το θέμα περισσότερο και χαίρομαι και που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ήδη ε, έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται και να βελτιώνει τις παρούσες σχέσεις. Το, η παρούσα συμφωνία πλαίσιο ε, ολοκληρώνεται το 2020. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει αρκετός χρόνος ε, ώστε να συζητηθούν τα επόμενα βήματα. Και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να συνεχιστεί η συζήτηση είτε σε αυτό είτε σε οποιοδήποτε άλλο βήμα για το θέμα αυτό. κύριος ε, Μπερμοντό. Ναι, ευχαριστώ. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ως τμήμα του σχεδίου δράσης ε, προβλέπουμε ε, έναν ακόμα έλεγχο επιδόσεων το 2020 για όλες τις δράσεις ε, των πολυμέσων, όχι μόνο το Euronews. Και εδώ δεν ασχολούμαστε μόνο με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, αλλά έχουμε και δίκτυα ε, data-driven που κινούνται με βάση δεδομένα. Ε, Επίση, ε, δεν περιμένουμε παθητικά να αναλάβει η καθήκοντα η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συναντιόμαστε με ενδιαφερομένου που μπορεί να ενδιαφέρονται για ευρωπαϊκέ μεταδόσει για να μπορέσουμε να παρέχουμε και εναλλακτικέ λύσει. Θα καταρτήσουμε ένα κατάλογο με τις διάφορες εναλλακτικέ λύσει. Θα δούμε τι υπολογισμό θα έχουμε τι κόστος ε, θα υπάρχει για τη ε, σημαντική μείωση ε, της χρηματοδότησης, για παράδειγμα, του Euronews ή να επιλέξουμε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο και θα επανέλθουμε. Θα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Κοσλόφς για την δουλειά που έκανα και για αυτά τα οποία μας δώσατε για να σκεφτούμε και τον συνόλφο της ε, Κομισιόν. Να ευχαριστήσω και σας ε, για την συζήτηση. Νομίζω το θέμα θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Ε, ευχαριστώ και την Μόνικα Χόλμα, ως πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Υπερπολισμού. Θα μας απασχολήσει οπωσδήποτε το θέμα αυτό για λίγο καιρό ακόμα και θα καταλήξουμε νομίζω σε μια λογική λύση. Οπότε σας ευχαριστώ και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, κανονισμός κατεξιοδότηση για την αναθεώρηση του κανονισμού 1295 του 2013 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών ε, δικτών ε, στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη από την Κομισιόν. Έχουμε καλέσει σήμερα την Κομισιόν για να κάνει αυτήν την παρουσίαση. Ε, να σας παρακαλέσω λίγη ησυχία. Έχουμε καθυστερήσει. Σας παρακαλώ λοιπόν αν θέλετε να φύγετε από την αίθουσα κάντε το ήσυχα. Παρακαλώ λοιπόν να συνεχίσετε. Ε, ε, βγείτε από την αίθουσα άμα θέλετε να μιλήσετε για να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Οπωσδήποτε θα θυμάστε τις διάφορες συζητήσεις για την ανάγκη αξιολόγησης ε, ποιοτικών δικτών. Η Κομισιόν οπωσδήποτε ε, ξεκίνησε την διαδικασία αυτή για την πράξη κατεξοδότηση. λόγω της ε, προεκλογικής περίοδου όμως δεν μπόρεσε να την διαβάσει το Κοινοβούλιο τώρα το λάβαμε στις 18 Ιουλίου δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά γιατί ακολούσαν οι διακοπές. Η προθεσμία για το Κοινοβούλιο και Συμβούλιο είναι 18 ε, Σεπτεμβρίου, αν είναι να υπάρξει κάποια αντίρρηση. Οπότε θα πρέπει να οριστούν οι συγητές και σκιώδες συγητές ε, και ίσως να υπάρξει μια παράταση της ε, προθεσμίας για να υπάρξει η δυνατότητα να ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Ενημέρωσα λοιπόν σχετικό την Κομισιόν και η νέα προθεσμία για το Κοινοβούλιο είναι 18 Νοεμβρίου, οπότε έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο αλλά θα μπορούσαμε να ε, εισαγάγουμε μια δική μας εσωτερική προθεσμία. Εάν κάποιος λοιπόν έχει κάποια αντίρρηση μπορεί να στείλει ένα email στην γραμματεία και σε μένα. και μια τροπολογία για την απόρριψη στα αγγλικά μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου στις 12 για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Οκτώβριο και να τηρηθεί η προθεσμία του Νοεμβρίου. Εάν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, τότε δεν χρειάζεται να ληφθούν άλλα μέτρα πριν από τις 18 Νοεμβρίου. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν για 10 λεπτά για να μας κάνει μια γενική εισαγωγή και μετά μπορούν οι βουλευτές να θέσουν ερωτήσεις. Έχουμε τον κύριο Ντελγκάδο και τον κύριο Ντόσον για την Κομισιόν. Ποιος θα μιλήσει πρώτος, ο κύριος Ντελγκάδο. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Να σας παρουσιάσω λίγο το πλαίσιο της δουλειάς μας. Ε, στη, βασική, ε, στη νομική βάση του Creative Bureau έχουμε ε, ένα σύνολο δικτών, αρκετά σημαντικό, αλλά η αξιολόγηση ήταν αρκετά θετική για το πρόγραμμα ΜΕΝ, αλλά υπήρχαν αρκετοί περιορισμοί για τους παρόντες δείκτες. Ο κανονισμός λοιπόν αυτό κατά εξουσιοδότηση θέλει να συμπληρώσει, γιατί επιτρέπεται μόνο ο κανονισμού κατά εξουσιοδότηση να συμπληρώσουμε τους δείκτε για να καλύψουμε αυτού τους περιορισμού. Υπάρχει μια ιστορική διαδικασία για την προετοιμασία της ε, πράξης κατεξουσιοδότησης και το Δεκέμβριο του 2018 συζητήσαμε με του εμπειρογνώμονε που είχαν ορίσει τα κράτη-μέλη βάσει της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ε, είχε προσκληθεί και η Γραμματεία της Επιτροπής Πολιτισμού ως παρατηρητής. Μετά έγινε διοργα... διπηρεσιακή ε, διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ έχουμε την πρόταση η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα όλων αυτών των εσωτερικών και εξωτερικών συζητήσεων. Οι δείκτες λοιπόν που προτείνεται είναι σε τέσσερις ομάδες διαρθρωμένη ε, που βλέπετε στο άρθρο 1 του κανονισμού κατά εξουσιοδότηση. Υπάρχουν ε, ε, τέσσερις συμπληρωματικοί δείκτες που αφορούν το βασικό στόχο του προγράμματος και αυτοί συνήθως είναι προδιαγραφές ήδη υφιστάμενων δεκτών στην παρούσα νομική βάση. Μετά, στην παράγραφο 2 έχουμε πέντε συγκεκριμένους ε, δείκτες για τους στόχους, που είναι διευκρίνηση ε, των δικτών που διαθέτουμε ήδη, αλλά έχουμε και ποιοτικού δείκτες, ένα γενικό ποιοτικό δείκτη στο σημείο 4 και ε, συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες στο σημείο 5. Η τρίτη ομάδα αφορά τα μέσα ενημέρωσης και θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο Μάρτιν Ντάουσεν μετά για να ε, σας πει δύο λόγια παραπάνω για αυτά. Και ο τελευταίος, η τέταρτη ομάδα είναι για τον πολιτισμό μόνο και αφορούν το συγκεκριμένο στόχο του πολιτισμού. Έχουμε επιπλέον εννέα ειδικού δείκτες, αλλά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι και όπως βλέπετε προσπαθούμε να διευκρινίσουμε δείκτες οι οποίοι σχετίζονται με συγκεκριμένα μέτρα. Το βασικό στοιχείο εδώ είναι τα, τα συστήματα πληροφορικής. Ε, συνεργαστήκαμε με τους αδέλφους από τον εκτελεστικό οργανισμό για να συλλέξουμε τα ε, δεδομένα, να τα ανακτήσουμε και να τα κατηγοριοποιήσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να καθορίσει κάποιος ένα νέο δίκτυο, δεν είναι τόσο απλό. Και θα λάβετε σύντομα και μία παρουσίαση και για τους δείκτες που διαθέτουμε ήδη, αλλά και για τους νέους δείκτες μέσω μιας έκθεσης που θα εκπονεί τακτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι στις επόμενες εβδομάδες θα στείλουν στην Επιτροπή ε, την έκθεση παρακολούθησης για το 2018. Μπορώ να πω περισσότερα αν έχετε ερωτήσεις και τώρα να δώσω στο συνάδελφο, το λόγο, τον Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ, Ζωάου. Όπως είπε και ο συνάδελφος, θεωρούμε ότι οι δείκτες αυτοί αποτελούν μια ευκαιρία να εξηγήσουμε λίγο καλύτερα τα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα που έχει το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Και επομένως όταν καθορίστηκαν αυτοί οι δείκτες, η προσπάθειά μας επικεντρώθηκε σε μια πιο ε, οξία ματιά για το τι κάνει ακριβώς το πρόγραμμα, τι ε, προσέχουμε και πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα. Μέσω λοιπόν αυτών των δικτών προσπαθήσαμε να καλύψουμε τρεις διαστάσεις πιο συγκεκριμένα. Πρώτον, θα θέλαμε να καλύψουμε το το στόχο της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και της ανταγωνιστικότητας του οπτικοακουστικού τομέα. Επικεντρώμαστε δηλαδή πιο πολύ στα οπτικοακουστικά. Για παράδειγμα, ένας βασικός δείκτης για μας είναι η διεθνής ε, αναγνώριση ε, που ε, λαμβάνεται και υποστηρίζεται από τα μέσα ενημέρωσης. Σε μια διεθνή αγορά για μας αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη και για την εγγενή πολιτισμική αξία ενός έργου και την ποικιλομορφία ενός έργου, γιατί προέρχονται από διάφορες χώρες στην Ευρώπη και ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα σε μια αγορά, διότι η αναγνώριση από τους κριτικούς ορισμένες φορές προσελκύει την προσοχή ε, του ακροτηρίου ε, και των θεατών και φυσικά αυξάνει και τα έσοδα και τα κέρδη μιας ε, ταινίας. Ένας άλλος τρόπος για να αυξήσουμε την ποικιλομορφία και την ανταγωνιστικότητα είναι να υπάρχει ισότητα των φύλων, που όπως ξέρετε είναι κάτι το οποίο έχει έρθει στο προσκήνιο ιδιαίτερα στον οπτικοακουστικό τομέα προσφάτως. Για μα η ισότητα μεταξύ ανδρών και ε, γυναικών είναι θεμελιώδη αξία και είναι και στοιχείο ανταγωνιστικότητα, διότι θέλουμε να προσελκύσουμε ταλέντο από όλη την κοινωνία. Και φυσικά οι γυναίκε είναι το 50% τη κοινωνία μα και πρέπει να υπάρχει και ισορροπία. Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχόλησε την Επίτροπο και έχουμε δείκτες για να μετρήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στο πρόγραμμα. Ε, είναι ε, ευνοϊκά τα στοιχεία σε σχέση με τα ευρύτερα στοιχεία ε, ε, στον κλάδο. Το 50% για παράδειγμα στα προγράμματα εκπαίδευσης είναι γυναίκες, αλλά μπορούμε φυσικά να κάνουμε πολύ περισσότερα και θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε στενά. Δεύτερον, μια διάσταση που θέλουμε να καλύψουμε με τους δείκτες είναι να καλύπτουμε όλη την αλυσίδα αξίας του κλάδου. Για να μπορέσουμε να έχουμε εμείς κάποιο αντίκτυπο πρέπει να περάσουμε από την εκπαίδευση ε, στην ε, διανομή του έργου μας. Και οι δείκτες καλύπτουν όλες αυτές τις πτυχές. Και επίσης καλύπτουμε και τους διάφορους τρόπους με τους οποίους διατίθεται τα έργα στα διάφορα κανάλια, δηλαδή διάβλους μάλλον, στο σινεμά, στο κινηματογράφο, αλλά όχι μόνο εκεί, αλλά και στην τηλεόραση, αλλά όλο και περισσότερο και σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Καλύπτουμε όλα αυτά τα στοιχεία στους δείκτες μας και ε, κάθε σκέλος της αλυσίδας αξίας του κλάδου πρέπει να προσμετράται με διαφορετικό τρόπο, χρειαζόμαστε άλλα στοιχεία, επομένως επιλέξαμε προσεκτικά δείκτες μέσω των οποίων μπορούμε να έχουμε τις πηγές των δεδομένων ετησίως, ώστε να μπορούμε να κάνουμε ετήσια σύγκριση και να έχουμε και μία εικόνα των τάσεων που παρουσιάζονται κάθε χρόνο, που είναι πολύ σημαντικό. Τέλος, η άλλη διάσταση που περιλαμβάνουν οι δείκτες είναι ε, ένα σύνολο ποιοτικών και ποσοτικών δικτών. Ε, μέτρηση των τηλεθεατών, ε, των θεατών μάλλον εν γέννη και το μερίδιο αγοράς των ευρωπαϊκών έργων. Είναι ένας ποιοτικό ε, δείκτης για να αξιολογήσουμε και την υγεία του οπτικού ακουστικού μας τομέα. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα προσμετρήσουμε όλα. Ε, ε υπάρχουν κάποια σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να αξιολογήσουμε επίσης. Για παράδειγμα, καινοτομία. Ε, σε ποιο βαθμό έχουμε καινοτομία στα όσα γίνονται και αυτά καλύπτονται από τους δείκτες μας. Ε, κάτι τελευταίο εδώ, ε, το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, είναι κάτι που είπε και ο Ζωάο. Ε, κάναμε κάποιες δοκιμές για τους δείκτες αυτούς ήδη στην έκθεση παρακολούθησης η οποία συντάχθηκε για το 2018 και δημοσιεύθηκε προσφάτως στο διαδίκτυο και πιστεύουμε ότι η έκθεση παρακολούθηση δείχνει ότι αυτοί οι δείκτες ε, είναι και εύστοχοι και ουσιαστικοί. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα οπτικοακουστικά, το 2018 ε, μπορούμε να δούμε συγκεκριμένα πώς βοήθησαν τα μέσα για την διασυνοριακή κυκλοφορία. Πάνω από 400 νέες ταινίε ε, ε, έγιναν, που είναι το 25% της ετήσιας ευρωπαϊκής παραγωγής ταινιών. Επίσης, Είχαμε πάνω από 500 ε, πρεμιέρες ταινιών ε, διασυνοριακά. Και από τα στοιχεία που μας έδωσε το Ευρωπαϊκό Οπτικό Ακουστικό Παρατηρητήριο, το οποίο παρακολουθεί την αγορά συνολικά, αυτό δείχνει ότι έχουμε μια αύξηση της διασυνοριακής κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι έχουμε θετικό αντίκτυπο των μέσων. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τα έγγραφα. Ε, υπάρχουν ε, όλα τα έγγραφα της συνεδρίασης ε, στον τόπο της Επιτροπής και στο, μπορείτε να τα βρείτε στο e-committee, αλλά νομίζω ότι όλοι τα έχετε λάβει. Ο κύριος Φραγκόφσκι και ο κύριος Μοχάματ είναι οι δύο συντονιστές που είναι παρόντες αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ χρήσιμο για μας ότι ξεκινάει ο διάλογος για το Creative Europe και είναι σημαντικό να υπάρχουν ποιοτικοί δείκτες για να μπορεί κανείς να μετρήσει την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων. Όσον αφορά λοιπόν τους δείκτες που έχουμε, οι πιο πολύ είναι ποσοτικοί. Για τους ποιοτικούς δείκτες, πώς μπορείτε να μετρήσετε την πολυμορφία, την πολιτιστική και την προστιθέμενη αξία. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Έχετε τον κατάλογο και τα έχετε στο έγγραφο όλα αυτά. Έχουμε δείκτες ποιοτικούς, άρθρο 1, 2, 4 όσον αφορά την καινοτομία, την τεχνολογία και την ποιοτική αξιολόγηση. Πρέπει κανείς βεβαίως να είναι αρκετά ανοιχτός όσον αφορά τον ορισμό του ποιοτικού. Προσπαθούμε, αν θέλετε, να αξιολογήσουμε τις επιτυχίες. Τι είναι όμως μια επιτυχημένη, ε, ένα επιτυχημένο τέτοιο εγχείρημα. περίπου το 60% των προγραμμάτων, αν θέλετε, χρηματοδοτείται. Είμαστε απαιτητικοί από την αρχή. Εφαρμόζουμε πολύ ε, ποιοτικά κριτήρια και η αξιολόγηση που γίνεται ουσιαστικά στοχεύει να εντοπίσουμε αυτά τα επιτυχημένα σενάρια. Ο κύριος Ντόσον. Θέλω να συμπληρώσω αυτό που είπε ο συνάδελφος αυτές οι κατεξουδότητες πράξη αξιολογούν τα υπάρχοντα, τα σημερινά προγράμματα μέχρι το 2020. Πρόκειται για μια μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση για το 2017. Όλα τα νέα προγράμματα θα αξιολογηθούν βάσει των νέων προτεραιοτήτων και θα υπάρξει μια νέα σειρά δικτών. Πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές, αν θέλετε, διαδικασίες. Μιλήσατε για τις ποιοτικού δείκτες. Κοιτάμε, παραδείγματο χάρη, την καινοτομία. Όσον αφορά την καινοτομία, λοιπόν, υπάρχει το καλλιτεχνικό, υπάρχει το επιχειρηματικό κομμάτι και βεβαίως αυτό της ψυχαγωγίας. Και προσπαθούμε να αναλύσουμε όλες αυτές τις συνιστώσεις στα υπάρχοντα τουλάχιστον προγράμματα. Και έχουμε ένα συνεχή διάλογο με τα εμπλεκόμενα μέρη και έχουμε και τον εξειδικευμένο τύπο, διαβάζουμε τις κριτικές και τις αναλύσεις που υπάρχουν για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μοχάμαντ δεν είναι όμως στην αίθουσα. Θα ήθελα εγώ να κάνω μία ερώτηση όσον αφορά τους δείκτες ποσοτικούς και ποιοτικούς. Η επιλογή, όπως ε, είπατε, των προγραμμάτων. Οι δείκτες αυτοί είναι γνωστοί, είναι δημόσιοι και ουσιαστικά αφορούν και τους ε, δημιουργούς οι δημιουργοί γνωρίζουν τους δείκτες βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν τα προγράμματά τους. Αυτά είναι δημόσια. Είναι εσωτερική διαδικασία δηλαδή αυτή ή είναι και εξωτερική δημόσια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν είναι εσωτερικό το έγγραφο και έχουμε και μετά από την σύμφωνη γνώμη ούτως ή άλλως ε, του Κοινοβουλίου θα δημοσιευτεί. Κατόπιν, όπως ε, ανέφεραν οι συναδελφοί μου, η Κομισιόν προβλέπει να δημοσιεύει κάθε χρόνο μία έκθεση η οποία θα βασίζεται στους δείκτες αυτούς που υπάρχουν στην νομική βάση και τους νέους που θα καθοριστούν από την πράξη κατεξουσιοδότηση συλλέγουμε δεδομένα σε πολλές φάσεις, ε, σε πολλά επίπεδα. Στο επίπεδο των αιτήσεων, όταν οι αιτούντες ορίζουν ποιοι είναι οι στόχοι του έργου, αλλά επίσης συλλέγουμε και δεδομένα την στιγμή της εφαρμογής και όταν κλείσει το έργο. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό μεταξύ της πρώτης συλλογής ε, δεδομένων ε, όταν γίνονται οι αιτήσει και 2-3-4 χρόνια μερικές φορές όταν ολοκληρωθεί το έργο και βεβαίω τα βασικά δεδομένα θα είναι τα δεδομένα ενός ολοκληρωμένου έργου γιατί καμιά φορά το έργο είναι απλά μια πρόθεση και όχι συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν πολύπλοκο μηχανισμό για να διορθώσουμε τα δεδομένα όταν οριστικοποιηθεί το έργο. Αυτό είναι κάπως ε, διαφορετικό από τα κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια επιλογής ε, είναι δημόσια. Οι ετούντες ε, ξέρουν ε, ποια είναι. Βεβαίως υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του αποτελέσματος και της επιλογής των έργων, αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει για κάθε έργο, οι ενδιαφερόμενοι θα γνωρίζουν από την έκθεση παρακολούθησης που θα είναι δημόσια ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία που προκύπτουν από το πρόγραμμα και τι σημασία έχουν. Ευχαριστώ. Έχετε κάποιες ερωτήσεις για την διαδικασία, για την ουσία. Όχι, οπότε σας ευχαριστώ για τις ε, εξηγήσει σα. Α, η κυρία Μπάντινγκ. Ναι, ναι, θέλω να πω κάτι επί τη διαδικασία. Ζητάτε συγκεκριμένα σχόλια σε μια συγκεκριμένη πράξη. Με συγχωρείτε, ασκώ κριτική και στην Επιτροπή και σε εσά, αλλά το όνομα εδώ πέρα στην ημερήσια διάταξη δεν είναι το ίδιο με το έγγραφο. Το έγγραφο αναφέρεται στην Δημιουργική Ευρώπη, αλλά όχι στον τίτλο του εγγράφου. Οπότε κάποιοι από εμά δεν το φέρουμε. Εγώ δεν είχα καταλάβει δηλαδή γιατί είμαι καινούρια. Δεν κατάλαβα ότι αυτό το έγγραφο αφορούσε αυτήν τη συνεδρίαση. Οπότε δεν κατάλαβα τίποτα γιατί δεν τα έχω διαβάσει. Δεν είναι κανένα μεγάλο έγγραφο. Θα ήθελα να σα παρακαλέσω στο μέλλον να τυπώνετε μερικά αντίγραφα και να τα φέρνετε εδώ. Γιατί όταν γίνεται μια λεπτομερή συζήτηση βοηθούν τα τυπωμένα αντίγραφα. Αν θέλετε να τα τυπώσω εγώ να τα τυπώσω αλλά βάλτε το όνομα στην ημερήσια διάταξη, στο, το όνομα του εγγράφου που είναι εκεί στο σετ. Με συγχωρείτε, δουλεύω στον δημιουργικό κλάδο ε, ως ελεύθερη επαγγελματία για μικρές εταιρείε. Ε, έχω εργαστεί και για το BBC για 30 χρόνια. Αλλά δεν έχω τίποτα να πω σήμερα και σβήνει το μικρόφωνο του Γιατί δεν είχα προετοιμαστεί. Αυτό δεν είναι θέμα της ε, Κομισιόν, λέει η Πρόεδρος, είναι θέμα της Γραμματείας. Κανονικά πρέπει να το είχατε στείλει και την ε, πράξη κατεξιοδότηση. Εγώ το είχα δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί δεν έγινε. Θα, το δούμε, θα το δούμε. Οπότε στο μέλλον δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Κανονικά όλοι λαμβάνουν ε, το έγγραφο. Ε, κοιτάξτε, δεν ε, τυπώνουμε αντίγραφα εδώ πέρα γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοί τα θέλουν ε, και λίγες μέρες πριν, όχι μόνο εντός της αίθουσας. Θα δούμε τώρα αν έγινε κάποιο λάθος όταν τα έστειλαν. Αλλιώς σας προτείνω πάντα να κοιτάτε τα email της Επιτροπής. Καμιά φορά, δεν ξέρω, μπορεί να τα στείλανε στις διακοπές. Μπορεί να έγινε και αυτό. Ε, δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Ε, έχουμε τώρα επί Η προθεσμία είναι μέχρι τον μέχρι τις 12 ε, Σεπτεμβρίου 12 η ώρα. Αν θέλετε να απορρίψετε την πράξη κατεξιοδότηση, στείλτε τις παρατηρήσεις σας στα αγγλικά, αλλιώς ε, θα περάσει. Αυτά. 12 Σεπτεμβρίου, 12 η ώρα λοιπόν. Ευχαριστώ. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης. Η επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 3 η ώρα και Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 9 μέχρι το απόγευμα όλη μέρα. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι οι συντονιστές να παραμείνουν. Παρακαλώ, ναι. Κύριε Νίνας, να με συγχωρείτε που σας διακόπτω. συγγνώμη, επειδή προσπαθώ να σχηματίσω μια διακομματική ομάδα για τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες. Θα περιμένω. Όσοι θέλουν, παρακαλώ. Όσοι δεν θέλουν να φύγουν. Ναι, και χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο. Ναι, θα ήθελα να επισημάνω ακριβώς ε, ότι υπάρχει μια διακομματική ομάδα για τα κοινωνικά δικαιώματα των δημιουργών. Όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Υπάρχει και η ομάδα για τον κλάδο τον πολιτισμικό και νομίζω μίλησα και με τον συνάδελφο εκεί και μου είπε καλό να υπάρχουν και οι δύο πλευρές του νομίσματος. αν ενδιαφέρεστε λοιπόν θα περιμένω έξω από την αίθουσα. Και θα το στείλω και το βράδυ σε όλους τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές, αλλά ήθελα να το πω πρώτα στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ωραία πρωτοβουλία. sorry to stay here in the room so that we can follow up with the coordinators meeting. Παρακαλώ να παραμείνετε στην